του κυρίου Γκουαλτιέρη σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη-μέλη με νόμισμα το ευρώ. Υπάρχουν δύο συγγητές και ζήτησαν και οι δύο για το λόγο, ο κύριος Μπροκ και ο κύριος Γκουαλτιέρη. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα μακράς διαδικασίας συζητήσεων με το Συμβούλιο. Ο κύριος Μπροκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι αναγκαίος ώστε μακροπρόθεσμα να υπάρξει η νομική ασφάλεια που θα διασφαλιστεί και θα εκφράζεται αλληλεγγύη για χώρε που θα έχουν προβλήματα, αλληλεγγύη που θα διασφαλίσετε, θα διασφαλίσετε το ευρώ στη σταθερότητά του αλλά και τα αναγκαία θεσμικά όργανα. Και τα θέματα ανάπτυξη θα μπορούν από κοινού έτσι να αποσαφινιστούν. Αυτό μπορούσε μόνο με μια απλουστευμένη διαδικασία να λειτουργήσει. Απλουστευμένη τροποποίηση τη συνθήκη λόγω του χρόνου που μια κανονική διαδικασία θα απαιτούσε, που θα ήταν πολύ μεγαλύτερο, ε, και για να αποφύγουμε δημοψήφισμα στα κράτη-μέλη. Το Κοινοβούλιο όμω λέγει ότι αυτό δεν θα πρέπει να είναι μια τακτική συνήθι διαδικασία. Διότι εδώ θα έπρεπε κανονικά μια αλλαγή συνθήκη να ε, είχε ακολουθηθεί. Οι αρχικέ ε, προποθέσει ήταν τέτοιε που ήταν μια καθαρά διακυβερνητική προσέγγιση, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαδραμάτιζε ρόλο, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα όμω μπορούμε να σα ότι με βάση τι διαπραγματεύσει που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο τη ομάδα τη Ευρωζώνη, ότι σχεδόν σε όλα τα θέματα όπου πρόκειτο για την εξέταση προτάσεων βάσει λήψη απόφαση και τα συναφή, το πλαίσιο δηλαδή που έπρεπε να καθοριστεί για την πρόταση ενός κανονισμού ώστε σε μια ενωσιακή διαδικασία να ρυθμιστούν αυτά, ώστε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο Υπουργών να, να, γίνουν, να έχουν γίνει αυτά δεκτά και τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται σε αυτή τη διαδικασία να διαδραματίσει το ρόλο του. Και για αυτούς όλους τους λόγους είμαστε σε σχέση με αυτή την εκκίνηση, η γραμμή αφετηρία, σα το πω έτσι, δεν είμαστε όλοι απόλυτα ικανοποιημένοι, αλλά θα πρέπει αυτό το πλαίσιο να το χρησιμοποιήσουμε όπω ε, στο παρελθόν είχε ε, ξεκινήσει μια τέτοια προσέγγιση, ώστε να καταλήξουμε σε μια ενωσιακή διαδικασία, κοινοτική διαδικασία. Και γι' αυτό μπορούμε να σα προτείνουμε σήμερα αυτή η διαδικασία τροποποίηση ε, να εγκριθεί σε σχέση με το Συμβούλιο από πλευρά μα. Και έχουμε και αντίστοιχε τροποποίησει τροπολογίες ομόθυμα σε σχέση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων όπως έχουν προταθεί αυτά και πρέπει η δική μας ερμηνεία να διασφαλίσουμε ώστε με επιστολή του Προέδρου της Ομάδας Ευρωζώνης του Επιτρόπου Αρμοδίου για τα νομισματικά θέματα καθώς επίσης και με επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μπορέσουν αυτά να διασφαλιστούν. Αυτά θα είναι μια αξιόπιστη βάση πιστεύω ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε ως Ευρωκοινοβούλιο και με αυτόν τον τρόπο το ευρώ το οποίο είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη να διασφαλιστεί από κοινού και να μπορέσει να μετεξελιχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφο Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Λοιπόν, η έκθεση που καλούμεθα να ψηφίσουμε και όσον αφορά τι επιφυλάξει για να γίνει αναθεώρηση τη συνθήκη όσον αφορά το δικαιωματικό χαρακτήρα του μηχανισμού, παραμένουν ε, σαν θέσει, αλλά ταυτόχρονα εμεί προτείνουμε μια γνωμοδότηση που είναι θετική, διότι όπω εξήγησε και ο Έλμαρ Μπροκ, οι διαπραγματεύσει που διεξήχθησαν μα επέτρεψαν να πετύχουμε σημαντικού στόχου που αφορούν πάνω απ' όλα το γεγονός ότι οι αιρεσιμότητε που συνδέονται με τις ενισχύσεις καθορίζονται από έναν κανονισμό, δηλαδή μέσα μια διαδικασία συναπόφασης. Άρα είναι σωστό να τοποθετηθούμε θετικά επ' αυτού και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολλού συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι, ήταν προνόμιό μου να συνεργαστώ με τον Ροκ. Ήταν χρησιμότατε οι συμβουλέ του Έντζο Μπυρίλο και η δουλειά που έκαναν οι δύο εισηγητέ τη Επιτροπή ΕΚΟΝ, ε, Σικλούν και Γκοζέ, οι σκιώδε Νταφ, Χέφνερ και οι συντονιστέ των ομάδων βεβαίω και οι πρόεδροι των ομάδων που μα έδωσαν σημαντική πολιτική υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα σε σχέση με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου να αναφέρω ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ψηφοφορία. Ευχαριστώ για την παρουσία σας λοιπόν σε μια τόσο σημαντική στιγμή. Κυρίε και κύριοι, τώρα θα προχωρήσουμε στη συνέχεια και θα ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τροπολογία 27 κατά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 16 και τροπολογία 28 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Έχουμε συμβαστικές τροπολογίες 38, 39 και 40 της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής. Όσοι αυτές οι τροπολογίες είναι αποδεκτές, έχουν μεταφραστεί και είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σα ρωτήσω, υπάρχουν κάποιε ενστάσει, κάποιε αντιρρήσει για την ψήφιση. Δεν υπάρχουν. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτέ τι τρει τροπολογίε, συμβασικέ τροπολογίε, 38, 39 και 40. Είναι ονομαστική, με ονομαστική κλίση η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλε και όλοι. τέλο ψηφοφορία. Έγινε, έγιναν δεκτές ε, οι τροπολογίες αυτές. Τροπολογίες 30 και 19 καταπίπτουν. Εσείς διαδικαστικό, παρακαλώ. Δεν δουλεύει το μηχάνημά μου της ψηφοφορίας. Ναι, θα σε ευχαριστώ συνάδελφε. Μάλιστα. Τώρα θα ελέγξουμε την 463. Θα ελέγξουμε την 463. Τώρα, η τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 33. Αυτή όμως έχει αποσυρθεί από τον κύριο Γκουαλτιέρη. Εντάξει. Και έτσι ο εισηγητή Γκουαρτιέρη έχει αποσύρει την τροπολογία 33. Δεν θα την ψηφίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 34. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η τροπολογία 35 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε η τροπολογία 36 με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε και αυτή. Η τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 32. Η τροπολογία 24. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβαστική τροπολογία 37 από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις ή ενστάσεις να ψηφιστεί αυτή η συμβαστική τροπολογία δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ψηφίζουμε συμβαστική τροπολογία 37 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ ψήφισατε όλοι πέρας ψηφοφορίας δεκτή η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 7 και η τροπολογία 26 ταυτόσιμες ψηφίζουμε υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν η τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση νομοθετική πρόταση ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε στο σύνολό της με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που συνεργάστηκαν ώστε να μπορέσει να επιτεθεί αυτή η έκθεση, να συνταχθεί αυτή η έκθεση. Και περνάμε στη συνέχεια στο επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξή μας. Κυρίες και κύριοι, είναι το θέμα των επεξηγήσεων ψήφου. Επεξηγήσεις ψήφου που μπορούν να γίνουν όμως αύριο. Δεν θα έχουμε σήμερα επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ να μην δώσετε σήμερα επεξηγήσεις ψήφου. Έγινε κατανοητό.